Δεν θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε αυτόν τον κατάλογο γιατί θεωρούμε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Ο πλήρης κατάλογος όμως θα συμπεριληφθεί στα αρχεία, θα μείνει λοιπόν στα αρχεία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για να μπορεί να τα βρει όποιος θέλει ε, την διεθνή λογοδοσία σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Για τις ε, πολιτικές αρχές τώρα, υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο ελέγχου των πράξεών τους. Ούτε υπάρχει ένδειξη ότι συμμετείχαν ε, στον προγραμματισμό ή την υλοποίηση των ε, ε, δράσεων ασφαλείας ή συμμετείχαν στο ευρύτερο οικοδόμημα. Ωστόσο, μετά τις, τα όσα συνέβησαν τον Αύγουστο του 2017, τους έχουμε λάβει υπόψη εκφράζουμε την απογοήτευσή μας στο το γεγονό ότι η Αν δεν έχει ε, καταβάλει κάθε ε, προσπάθεια για να καταδικάσει αυτές τις εξελίξεις ε, στο κράτος Ρακάιν. Ελπίζουμε η διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση όχι μόνο για να δικαιωθούν τα θύματα, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε, σε απίστευτη κατάσταση, αλλά και για να αποτρέψουμε μελλοντικές αποτρόπες πράξεις. Ο κύριος Συντότη τώρα θα μιλήσει για το πλαίσιο που αφορά τη λογοδοσία. Έκανε λόγο για το μέλλον. Η έκθεση που παραδώσαμε αυτή την εβδομάδα και θα έχουμε και συμπληρωματική στο τέλος Σεπτεμβρίου κάνει αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Η λογοδοσία έχει να κάνει με το παρελθόν και με τον προσαχθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για ε, ε κάποια από τα πιο δεχθεί εγκλήματα. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου. Στην περίπτωση του Ρακάιν, γενοκτονή, στην περίπτωση του Ρακάιν, τα πιο σοβαρά εγκλήματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν να να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική λογοδοσία στην ε, Μιαμάρ. Εδώ και 50 χρόνια δεν έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη Μιαμάρ. Έχουν γίνει πολλέ εσωτερικέ έρευνε χωρίς κανένα αποτέλεσμα τα τελευταία 8 χρόνια. Η μόνη δυνατότητα αποτελεσματική λογοδοσία είναι μέσω του διεθνού συστήματο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προτείνει έναν διεθνή δικαστικό μηχανισμό για να προσαχθούν εγκληματίες, ε, ενδεχόμενοι εγκληματίες για να αποφαστεί να θόει η ένοχη. Εννέα έχουμε κατονομάσει που θα πρέπει να διερευθούν και να προσαχθούν. Είναι θέμα ε, δικαστηρίου να αποφασίσει για την αθότητα την ενοχή τους. Έχουμε κάνει κάποια προπαρασκευαστικά βήματα για να λάβουν χώρα οι έρευνες και οι προσαγωγές και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η παρακολούθηση και η σύνταξη εκθέσεων έχει να κάνει με το παρόν. Είναι ιστορικά αυτά που έχουμε ανακαλύψει, αλλά συνεχίζουν να συμβαίνουν Φυσικά υπάρχει η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία δεν έχει τελειώσει αλλά συνεχίζεται και δεν υπάρχουν προοπτικές να σταματήσει. Ακόμα και φέτος το κράτος του Ρακάιν με το τρέχον καθεστώς αποχωρήσεων προς τον Μπαγκλαντές θα υπάρξουν άλλοι 20.000 ρογγίχια που θα περάσουν τα σύνορα. Δεν σταματάει λοιπόν ε, ούτε στο κατσίν ούτε στο τσάν. στο τελευταίους έξι μήνες εστιάσαμε στο Ρακάιν. Ο πόλεμος έχει εντικοποιηθεί στο Κατσίν και στο Τσάν. Χρειάζεται στενότερη παρακολούθηση ώστε αυτά που συμβαίνουν να ε, παρουσιαστούν στον κόσμο. Μιλάμε όμως και για το μέλλον. Η συνδική κυριαρχία τα τελευταία 50 χρόνια συνδέεται με μορισία. Πολύ μικρός αριθμός στρατιωτών έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Ο στρατός ως θεσμός και η στρατηγοί είχαν πλήρη ατιμορρυσία για μισό αιώνα. Πότε θα σταματήσει η και αν δεν συμβεί αυτό, αν δεν σταματήσει αυτή η ατιμορρησία και δεν αποδοθούν, αποδοθούν οι ευθύνε, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση στην ε, Μιαμάρ. Θα συνεχιστούν τα εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ε, ρόλο να παίξει. Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζει. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια μέχρι στιγμής είναι σχεδόν ανυπαρκτή. Αυτοί που έχουν κατονομαστεί και θα πρέπει να προσαχθούν, θα πρέπει ε, να υποστούν κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε ταχαίως, αλλά πρέπει να προσταθούν με αυτά τα στον κατάλογο. Θα πρέπει επίσης ο στρατός του Μιαμάρ ε, να αποδυναμωθεί. Θα πρέπει μια προτεραιότητα να είναι η αστυνομία να μην αποτελεί πλέον κομμάτι του στρατού, όχι μόνο για να διορθώσουμε το παρελθόν, αλλά για να σταματήσουμε κάτι τέτοιο από το να ξανασυμβεί. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των κρατών μελών και των διεθνών θεσμών, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις ομιλητές και σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας για την ερευνητική αποστολή. Στο σημείο 12 λέει ανταλλαγή απόψεων ε, με τους βουλευτές. Θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές λοιπόν. Έχω στον καταλογό μου. Mr. Panzeri, Ms. Gomez, Ms. Gill, Mr. Khan, Mr. Leitz, Mr. Bashir, Mr. Van Orden, Mr. and Ms. Lochbieler. Did I miss anyone? Ξέχασα κανέναν. Σε με Τζέφρι. Έχουμε περίπου 25 λεπτά στη διάθεσή μας. Ένα-δύο λεπτά ίσως ε, θα μπορούσατε να πάρετε το λόγο και κατόπιν θα απαντήσουν οι προσκεκλημένοι. Ο κύριος Παντζέρη καταρχήν ως πρόεδρος της Επιτροπής. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την πλευρά της ε, Επιτροπής μας ε, για το έργο σας ε, και μία αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επισκέφθηκε τη Μιερμάρ πριν κάποιους μήνες και καταρχήν περάσαμε από το Κοσβατζάρ και συνειδητοποίησε την κατάσταση. Η γενική εντύπωση που αποκομίσαμε είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή φάση στην ε, διαδικασία της δημοκρατικής μετάβασης. Υπάρχει συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και πραγματικά μας υπογοητεύει η στάση της Αγξουκή. Στο πλαίσιο αυτό οι βιοπραγίες κατά το Ροχίγια μας δείχνουν την πτυχή της πιο βυθιάς κρίσης που βιώνει η χώρα. Εμείς στις συναντήσεις που είχαμε για να συζητήσουμε ακριβώς αυτή την υπόθεση, ρωτήσαμε τέσσερα πράγματα που θέλω, ζητήσαμε τέσσερα πράγματα που θέλω να επαναλάβω. Δηλαδή, αυτό που ζήτησε ο Κόφι ε, να υπάρξει πραγματική παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα ε, και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο Ρακάιν. Επίσης, ε, να εφαρμοστεί η συμφωνία μεταξύ Μιανμάρ και Μπαγκλαμές προκειμένου να μπορούν να επιστρέψουν οι πρόσφυγες με την συμμετοχή και της υπετσαρμοστίας να αλλάξει ο νόμος του 1982 για την Ιθαγένεια για να ληχθεί το θέμα των απάτριδων και να δημιουργηθεί και μία Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή που θα αποδώσει την ευθύνη ε, για τα εγκλήματα. Βέβαια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ πιστεύω το έργο σας ε, θα χρησιμεύσει προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι τέσσερις στόχοι. Ευχαριστούμε κύριε Παντζιέρη. Τώρα το πρόεδρο, ο κύριος Λάνγκη έχει το λόγο που είναι πρόεδρος ε, της ε, αντιπροσωπείας για την Ασία. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου. Θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση. Η κατάσταση στη μία μα σε σχέση με τους Ροχίνγκια είναι πραγματικά δραματική. Παρόλε τις προσπάθειες να μειώσουμε την ισχύ του στρατού. Δεν το καταφέραμε. Μέχρι το 2012 υπήρχαν ε, μεγάλες κυρώσεις ενάντια εις Βαρτσελίτ. Το 2011 ε, έγινε λόγος για μεταρρύθμιση τεγματική. Στο μεταξύ, μάρα έγινε μια από τις φτωχότερες χώρες γιατί ε, ο στρατός συνέδεσε το νόμισμα με το δολάριο και χρησιμοποίησε τους φυσικούς πόρους αποκλειστικά, κάτι που δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Aung Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τελευταία συνομιλία ότι θα μπορούσατε να στραφείτε ενάντια του στρατού, αλλά αυτό θα οδηγούσε σε εμφυλίο πόλεμο. Θα μπορούσαν να νοθούν ε, επίσης οι κυρώσεις και η απαγόρευση εισόδου στη χώρα για να πετύχουμε κάτι. Τον επόμενο μήνα έχουμε σύνοδο. Το θέμα το Ροχίνγκια είναι στο επίκεντρο. Θα συμμετέχουν ε, ε, πιέζουν κοινοβούλια και από την περιοχή, από την Δονησία και από άλλες χώρες της περιοχής να επιτευχθεί βελτίωση της κατάστασης στη Μιαμάρ και να ε, τηρηθούν και να ληφθούν μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο Ισιάρ Τζέφρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για αυτή την ε, πολύ καλή έκθεση, για αυτή την ε, βαθιά τραγική κατάσταση που αφορά τους Ροχίνγκια. Για πολλά χρόνια ζητούσαμε δημοκρατική αλλαγή στη Μιανμάρ. Και αυτή είναι μια ακόμη τραγική εξέλιξη. Έχω δύο συγκεκριμένες ανησυχίες. Καταρχήν έχω μια ερώτηση. Έχουν υπάρξει καταγγελίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βιασμών που έγιναν ε, στους καταβλισμούς από άνδρες ε, Ροχίνγκια και θα ήθελα να ρωτήσω αν βρήκατε κάποιες αποδείξεις ε, γιατί αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και θα ήθελα να ξέρω αν το γνωρίζετε. Αλλά η συγκεκριμένη μου ανησυχία έχει να κάνει με την καταδίκη της Αγκ ε, δεδομένου ε, της αμφίσιμης θέσης της. Και ε, πραγματικά αναρωτιέμαι με την ικανότητά της να ελέγξει το στρατό στη Μιανμάρ. Μιλήσατε για το μέλλον. Θα πρότεινα ότι ένας ε, πόλος ελπίδας που έχουμε είναι μέσω της Αν Σαν Σουκί. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και προτείνω επομένως, ε, αντί να την υποσκάπτουμε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα καλύτερα ένστικτα σε αυτήν και να υποστηρίξουμε το ρόλο της, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω ποιος, ε, σε ποιον άλλο θα μπορεί να απευθύνει κανείς έκκληση στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, Τζέφρι. Από το Άλντε, ο κύριος Νάρτ. Ε, μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια αμφισημία εδώ γιατί η Ανσουκή είχε λάβει την υποστήριξη από όλη τη διεθνή κοινότητα όταν υφίστατο ε, ουσιαστικά πολύ μικρότερα δεινά από τους Ροχίνγκια. Και μπορώ να πω ότι ε, κύριος ο γενικός της ε, διευθυντής ε, ουσιαστικά απευθύνθηκε στον εισαγγελέα για να υπάρξει απέλαση προς τον Μπεγκλαντές. Τι είπε αυτό ο κυρίω και τι είπε η Πρωθυπουργό ότι το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία. Δηλαδή το ίδιο που θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε μοσταγή δικτάτορα σε σχέση με τα εγκλήματα που έγιναν. Σίγουρα στην σχιζοφρενική κατάσταση της Βερμανίας ε, η διαφορά μεταξύ της εξουσίας και της πραγματικής εξουσίας που την έχει ο στρατός είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει και μια ηθική αναγκαιότητα. Και στην περίπτωση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσει αυτά που έγιναν και σε σχέση με το βραβείο Σαχάροφ. Είναι εντελώς απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μην μιλά και να εξακολουθεί να μην αποσύρει το βραβείο Σαχάροφ από την Ανσουκή. Επομένως, αν μας ε, μένει ένα υπόλοιμα αξιοπρέπεια, το που πρέπει να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βρούμε μια φόρμουλα που δεν υπάρχει και που θα είναι ή ε, ε, να απορρίψουμε, να την απορρίψουμε την Ανσουκή και να τις αποσύρουμε το βραβείο Ζαχάρο. Διαφορετικά το μόνο που μας απομένει είναι υποκρισία. Μπίλερ, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την έκθεση. Εσείς συστήνετε είτε να παραπευθούν ε, οι στρατηγοί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή να συσταθεί ένας ε, διεθνής μηχανισμός λογοδοσίας. Εμείς στο ψήφισμά μας ως Κοινοβούλιο επίσης πιστεύουμε ότι αυτές οι στάσεις ε, είναι ορθές. Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα για να το πετύχουμε αυτό. Κύριε Συντότη είπατε ότι συστήνεται έναν διεθνή δικαστικό μηχανισμό. Ποια είναι η διαφορά ή μήπω είναι το ίδιο με αυτό που ζητά ειδικό απεσταλμένο του ΙΕ στη σε σχέση με τις ευθύνε ε, τη ε, αστική κυβέρνηση. Αναφέρατε πάρα πολλέ με στρατιωτικέ κυβέρνησεις ότι απέκρυψαν τις ε, βιοπραγίε, τις αποτρόπιες πράξεις, ότι η μη στρατιωτική κυβέρνηση συνεχίζει να παραπλανεί και ότι ουσιαστικά ε, προβαίνει και σε καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Οι αποδείξει που έχουμε πιστεύετε ότι είναι ε, τόσο ισχυρέ που θα μπορέσουν να σταθούν και στι διάφορε δικαστικέ διαδικασίες. Δεν μπόρεσα να διαβάσω το σύνολο της έκθεσης. Ε, αναφερθήκατε στο ρόλο κάποιων ε, ριζοσπαστικών βουδιστών μοναχών και στην ευθύνη που έχουν για αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καν για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι για αυτή την ε, έκθεση. Είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο ε, αυτό που γίνεται μέσω της διερευνητικής αποστολής, όμως ε, τώρα θα πρέπει να προβούμε σε έρευνες για την απαγγελία κατηγοριών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει για ένα ισχυρό ψήφισμα που να καλέσει το Συμβουλίο Ασφαλείας να παραπέμψει τη Μιανμάρ στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Έχω τρει ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν έναν εξάρτητο και μερόληπτο μηχανισμό. Δεύτερον, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αποτύχει να ε, υπερασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μήπω ε, θα πρέπει να γίνει μια έρευνα και για την εμπλοκή του ΟΗΕ στη Μιανμάρα από το 2011. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά. Και τρίτη ερώτηση, υπάρχει μεγάλη υποχρηματοδότηση και υπάρχει βάρος άχθος για τον Μπαγκλαντές αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους ε, Ροχίνγκια και την κοινότητα Ροχίνγκια, αλλά και την ε, κοινότητα υποδοχής τους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ροχίνγκια αλλά και την κοινότητα υποδοχής τους. Ευχαριστώ, κύριος Μπασίερ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση. Εγώ ήμουν εκεί πέρσι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο όταν είχαμε τη μαζική έξοδο και ήμουν μάρτυρας ε, της πυρπόληση στο χωριό. Η έκθεσή σας ε, ε, ε, σωστά επικεντρώνεται στα διάφορα φαινόμενα, Όμω, πού πάμε από εδώ και πέρα, ο ΙΕ θα παραπέμψει αυτό το θέμα στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Πιθανότητα θα τεθεί βέτο από την Κίνα. Και αν τεθεί βέτο από την Κίνα, τότε ε, μπορεί να πάει στην Γενική Συνέλευση και να ε, παρακάμψει το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η Μιανμάρ θα πρέπει να συνεργαστεί. Κάτι που δεν είναι και πολύ πιθανό. Ωστόσο, ξέρετε ότι πέρσι απευθύναμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια διεθνής σύνοδος κορφής μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να βρούμε ένα τρόπο επαναπατρισμού, να επαναπατριστούν οι Ροχίνγκια και να αποκατασταθούν τα δικαιώματά τους μια, και μια ανεξάρτητη έρευνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας να λάβει χώρα. Ποιε είναι οι απόψεις σας για μια διεθνή διάσκεψη ε, που θα μπορούσε να οργανωθεί από κοινού με τον ΟΗΑ για να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Έχω πάει πολλές φορές στον Μπαγκλαντές. Είναι ένα τεράστιο άχθος ε, σε μια χώρα σαν τον Μπαγκλαντές. Μήπω θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον Μπαγκλαντές ε, να δημιουργήσει ειδικέ οικονομικές ζώνες για τους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να ε, μπορούν να κερδίζουν ένα μεροκάματο και επίση να επενδύσουμε σε υποδομέ και στη Μιανμάρ και στον Μπαγκλαντές ε, για να μπορέσουν να επαληστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμας. Σας ευχαριστώ πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερως που σας ε, βλέπω εδώ μαζί μας. Κάποιος από εσάς σας ξέρω και από μια προηγούμενη ζωή. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση και για την συγκεκριμένη περιοχή και για τον κόσμο. Η έκθεσή σας είναι εξαιρετικά σημαντική. Και θα ήθελα να επισημάνω και την ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2015 στις εκλογές στη Μιανμάρ και είχαμε προειδοποιήσει, μπορώ με περηφάνεια να πω, ότι είχαμε προειδοποιήσει για τους κινδύνους ε, στην χώρα αυτή. Ε, υπήρξε προσπάθεια αποσιώπησης των όσων είχαμε να πούμε, αλλά δεν τα κατάφεραν. Εμείς προειδοποιήσαμε είδαμε και την ευθύνη των βουδιστών μοναχών, γιατί... Ε, προσπαθούν να διαδώσουν ε, τον πλέον ριζοσπαστικό ε, Ισλάμ, αλλά και την ευθύνη πολιτικών, όπως και η Ανσουσί, που μεταλείπει πρέπει να πω, και το είχαμε επισημάνει σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, γιατί και εμείς ήρθαμε σε επαφή με τους εκπροσώπους των Ροχίνγκια, που ήδη τότε, από τον Νοέμβριο του 2015, ανέφεραν ε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει αυτό που συνέβη τελικά. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, είναι το ερώτημα. Σίγουρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει λόγω και Ρουσίας και Κίνας. Αλλά εσείς βλέπετε κάποια δυνατότητα εφόσον 130 βουλευτές από χώρες της Ασίας υποστήριξαν με δήλωσή τους την έκθεσή σας και ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ε, να ε, προσάγει τους ηθήνοντες. Άκουσα αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι δεν γίνεται να λέμε ότι λόγω γεωστρατηγικών λόγων ή άλλων ότι ε, ξεχνάμε τα δικαιώματα, παρότι θα υπάρξουν τέτοιε προσπάθειε. Στην πράξη, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε έναν κατάλογο. Θα είναι αποτελεσματικός αυτός ο κατάλογος αν διαφύγουν οι ένοχοι της δικαιοσύνης. Σίγουρα θα υπάρξουν ένοχοι και εκτός της Μιανμάρ. Ευχαριστώ, Ανιλίτς, τώρα. Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Άννα θα είμαι πιο σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο πλευρό σας και εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Τι περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε κι εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός φορέας. Ε, παρακαλώ πείτε μας τι θεωρείτε ότι μπορεί και οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Είναι αγκαίο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους ε, τους προηγούμενους ομιλητές. Ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη η έκθεσή σας, ιδιαίτερα ανησυχητική επίσης. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ρόλο που βλέπετε να διαδραματίζει η διεθνή κοινότητα και ο ΙΕ. Λέτε ότι θα πρέπει ε, να βρεθούν στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών. Ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι αν θεωρούμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι μονόδρομος, όπως ανέφεραν κάποιοι εκεί έξω, ότι αυτή η στρατηγή θα πρέπει να προσαχθούν ενώπιον του ε, Διεθνούς ε, Δικαστηρίου. Η Μιανμάρ όμω δεν ε, εμπίπτει στη δικαιοδοσία του. Μπορεί να γίνει αυτό μέσω του Μπαγκλαντές. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το λύσουμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει ε, ένας οδικός χάρτης από την αναγνώριση της γενοκτονίας που είναι σαφής, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να φτάσουμε στην ειρήνη και τη συμφιλίωση, αλλά και για την αποκατάσταση των εκτοπιστέντων. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που θέλετε ε, από εδώ και πέρα, για να τα βάλουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο ε, στις εκθέσεις μας από εδώ και πέρα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αγγίλ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο τον λόγο. Ίσως λοιπόν μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο γίνεται σε περισσότερα ερωτήματα εντός 4-5 λεπτών έκαστος. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος, ε, πρώτα οι κυρίες, πρώτα οι Αστραλοί. Οι κυρίες προηγούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Είναι πολύ σημαντικά και για μας για να κατανοήσουμε αλλά και για την διεθνή κοινότητα για να βρει ε, τα επόμενα βήματά της μέσα στους επόμενους μήνες και έτη. Ένα λεπτό ζήτημα που θέσατε είναι ότι το Τατμαντόρ άνοιξε το 2011 και τώρα ξανακλίνει. Ήταν το πρώτο θύμα και είδαμε ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν πρέπει να συνδράβουμε τους αμάχους και τους πολίτες της Μιανμάρ, δίνοντάς τους την αλήθεια και μακροπρόθεσμα ελπίζουμε να λάμψει αλήθεια, παρότι μπορεί να τους λέει άλλα η κυβέρνησή τους. Θέλουμε λοιπόν να λάμψει αλήθεια και να κατανοήσει ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει στη ΜΜΑΡ. Κάτι άλλο για του καταβλισμού και την ε, σεξουαλική βία εκεί. Ναι, υπάρχει ε, σεξουαλική βία στου καταβλισμού και ενδοκογενειακή βία. και οι ΜΚΟ και οι γιατροί χωρίς σύνορα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Κάποιοι έχουν, ε, έχουν γίνει ανάδοχοι ορισμένων οικογενειών στους Η φύση, λοιπόν το ζήτημα, έχει αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό. Θέσατε μετά το ζήτημα της Ανσουκή. Στην έκθεσή μας ε, θέλαμε να διευκρινίσουμε και να καταστήσουμε ιδιαίτερα σαφές ποιος έχει την μείζωνα ευθύνη και ποιος ε, βρίσκεται σε ε, θέση να αποφασίζει, ποιος έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Ε, και αυτό είναι η στρατιωτική ηγεσία. Η Αν λοιπόν, με βάση τις συνταγματικές της εξουσίες, δεν βρίσκεται σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις ή καν να έχει γνώση στην αρχή του τι συνέβαινε. Αλλά στη συνέχεια, παρότι υπάρχει κάτι τέτοιο και παρότι ισχύει αυτό στη συνέχεια με το να παρεμποδίζει τις έρευνες και με το να διαδίδει ψευδή αφηγήματα και ούτω καθεξής, ε, έχει και εκείνη συνεισφέρει στις βιοπραγίες. Βέβαια, άλλοι είναι τα τέρατα με βάση τα στοιχεία που βρήκαμε εμείς. Επομένω, δεν ε, εκμεταλλεύτηκε την ε, θέση της, αλλά δεν, είναι, δεν υπάρχει εγκληματικός και δόλος, αν θέλετε, από ποινική άποψη. Μετά για τους βουδιστές μοναχούς που αναφέρατε. Εξετάσαμε μία ομάδα που τώρα έχει διαλυθεί και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έχει μακρά παράδοση ε, τέτοιων ακραίων βουδιστών μοναχών. Πάντα όμως το θέμα δεν είναι η ύπαρξη μιας ακραίας ε, ριζοσπαστικής ομάδας, αλλά πώς το κράτος ε, αντιμετωπίζει αυτές τις ομάδες. Το θέμα λοιπόν στη Μανμάρ είναι ότι το κράτος τους επέτρεψε να κάνουν ό,τι θέλουν. με πλήρη ατιμορρησία σε ό,τι αφορά την ρητορική μίσου, ε, τις ε, σειράξεις ε, χαμηλής κλίμακας. Δεν υπήρξε καμία αντιμετώπιση αυτού του εξτρεμισμού. Τώρα σε ένα βαθμό κάπως τους αντιμετωπίζουν, αλλά όχι αρκετά. και ο στρατός ε, κάπως παίζει με αυτή την ιδεολογία για να στηρίζει και να αυξάνεται, να γίνονται πιο δημοφιλείς. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, συγγνώμη, αλλά τελειώνει ο χρόνος. Επόμενος. Παρακαλώ, κύριο Σιντότη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αρκετά ερωτήματα αφορούσαν ε, την ποινική λογοδοσία. Θα σταθώ λοιπόν σε αυτό κατά βάση. Χρησιμοποίησαμε την ορολογία αυτή, διεθνή μηχανισμό ποινική λογοδοσία, γιατί το πιο σημαντικό για μα είναι να υπάρχει αυτή η διεθνή ποινική δικοδοσία. Και μετά το τι σημαίνει αυτό είναι δευτερεύον. Το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο έχει θεσπιστεί ακριβώ με αυτό το σκοπό. Γι' αυτό υπάρχει. Και είναι ο πλέον αρμόδιο φορέα. Όμω η Μιανμάρ δεν εμπίπτει στην δικαιοδοσία, ε, όπω αναφέρθηκε. Ε, υπάρχει μία υπόθεση ε, για το κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό μέσω Μπαγκλαντές. Αυτό ισχύει μόνο για τις απελάσεις προς το παρόν. Μπορεί να υπάρξει παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά Είπατε και εσείς ότι γνωρίζετε ε, τις δυσκολίες που υπάρχουν εκεί. Αλλά είναι εύλογο να περάσουν όλα αυτά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Μπορεί να γίνει και μέσω ειδικού δικαστηρίου. Ε, το Συμβούλιο Ασφαλής το έχει κάνει αυτό για τη Ρουάντα και για τη Γιουγκοσλαβία Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα εξετάσουμε. Η Ρωσία και η Κίνα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ίσως ε, άλλο δικαστήριο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει άλλα ζητήματα μετά θα μπορούσε να υπάρξει, ε, ε, να θεσπιστεί ειδικό δικαστήριο ε, μέσω συνθήκης. Και το ίδιο το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο μέσω συνθήκη είχε θεσπιστεί. Καλύπτει μια συγκεκριμένη γκάμα εγκλημάτων. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δικαστήριο. Και το σημαντικό είναι ότι τα εθνικά δικαστήρια ασκούν διεθνή δικαιοδοσία. Ε, και γι' αυτό κατονομάζουμε τους ηθήνοντες. Ούτως ώστε να γνωρίζουν οι ένοχοι ότι μπορούν να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οπουδήποτε κι αν πάνε, σε οποιαδήποτε χώρα. Αλλά αυτά τα επισημαίνουμε και στην έκθεσή μας. Το πιο σημαντικό είναι η λογοδοσία. Ο τρόπος και το μέσο ε, που θα επιτευχθεί η λογοδοσία είναι ένα σημαντικό αλλά δευτερεύον ζήτημα. Θα ήθελα, εν συντομία, να σταθώ στο ζήτημα της δημοκρατικής μετάβασης και να πω το εξής. Πράγματι, υπάρχει μια τέτοια δημοκρατική μετάβαση που λαμβάνει η χώρα στην Μιανμάρα. Αλλά από την αισιοδοξία μας έχουμε ε, υπερβάλλει στην ταχύτητα με την οποία ε, υλοποιείται αυτή η μετάβαση. Μόλις έχει ξεκινήσει λοιπόν στην ουσία αυτή η διαδικασία. Η Ντούρς είναι η καλύτερη δυνατότητα που έχει η Μιανμάρ, αλλά καμία από τις ε, κοινότητες και τις μειονότητες ε, της ε, Μιανμάρ και οποιοδήποτε πολιτικός φορέας δεν πρόκειται να ωφεληθεί από το να αποκρύπτει την πραγματικότητα και να συμμετέχει σε αυτή την συνωμοσία απόκρυψης της αλήθειας. Πρέπει να, κανείς λοιπόν να είναι ανοιχτός και διαφανής. Ευχαριστώ. Uh, uh, Να συμφωνήσουμε με την κυρία Γκομέζ. Έχουμε ένα μεγάλο άλμα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Κύριε Πρόεδρε, Ορθή η σειρά με την οποία μας αναθέσετε να μιλήσουμε. Να αποσαφηνίσω το λόγο που ήρθαμε εδώ στις Βρυξέλλες για δύο μέρες αρχικά για να ενημερώσουμε και από τους δύο και εγώ και οι δύο συναδελφοί μου να ευαισθητοποιήσουμε ως προς το πρόβλημα την κλίμακά του τη φύση, τα εγκλήματα και τη συνέχεια της κατάστασης. Έχουμε να κάνουμε με πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Συνεχίζεται η κατάσταση. Επίσης θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο να προσεγγίσουμε μια λήψη απόφαση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνθήκαμε με θεσμού, οργανισμού. Έχουμε μια συνάντηση στο Ινστιτούτο για Ασιατικές ε, Σπουδές για να συζητήσουμε για κάποια πιο ακαδημαϊκά θέματα ενδεχομένω, αλλά όμω ο στόχος είναι να καθορίσουμε την πορεία από εδώ και στο εξή. Ο ένας δρόμος έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο δεύτερος είναι με την ανθρωπιστική διάσταση και ο τρίτος δρόμος έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Είναι πολύ σκοτεινή εικόνα, θλιβερή στη Μιαμάρ. Όμως, παρόλα αυτά, ελπίζουμε ότι είναι κάτι που μπορεί να διευθυντηθεί. Η ερώτηση, τι μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο, είναι να συνεχίσει να ασκεί πίεση, να εφαρμόσει πίεση στο δικαστικό τομέα σε αυτά τα τρία μονοπάτια Έχουμε εντοπίσει τα ονόματα αυτών που πιστεύαμε ότι είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τα αποτρόπαια εγκλήματα από συλλογική ευθύνη περνάμε στην ατομική ενοχή. Θα πρέπει να αποκατασταθούν τα πράγματα, να αποκατασταθούν τα πράγματα, όχι να τιμωρηθεί το έθνος. Στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σε διεθνές επίπεδο είναι μια στιγμή που θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν δεν παρεμποδίσουμε την γενοκτονία θέτοντας σε ισχύ μηχανισμούς και η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ακριβώς αυτό, να πράξουμε αυτό όσον αφορά τα άμεσα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι πήγον να εστιάσουμε στην ανθρωπιστική διάσταση. Η κατάσταση των Ροχίνγκια στον Μπαγκλαντές χρήζει διεθνούς κινητοποίησης πόρων. Αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια σταθερή διαδικασία προσέγγιση της κυβέρνησης της Μιαμάρ, θα φτάσουμε ένα σημείο όπου θα υπάρξει μια α, συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας. Έτσι βλέπουμε το πρόβλημα και ε, αναμένουμε από εσάς να εγκριθεί το ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 18 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της ε, Διερευνητικής ε, Επιτροπής, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μας δώσετε. On behalf of our colleagues from των μέλλον τη Επιτροπή, να σας ευχαριστήσω που παρουσιάσετε τα πορίσματα της διευρυντική αποστολή. Πολύ σημαντικό το έργο σας και σα ευχόμαστε τα καλύτερα. Ελπίζουμε να έχετε δύο ενδιαφέρουσε μέρες ε, εδώ στις Βρυξέλλες. Σα ευχαριστούμε και πάλι που μας επισκεφτήκατε στην Επιτροπή.